είναι στο έλεος των λαθροδιακινητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κρύβονται μέσα σε κυβότια. Είναι ε, ε, άνθρωποι ε, που χρειάζονται την υποστήριξή μας. Επίσης, στη Σουηδία έχουμε παράνομο εμπόριο καυσίμων. Ήρθε λοιπόν ο, η στιγμή άμεσα να βάλουμε ένα τέλος σε όλα αυτά, αν θέλουμε πραγματικά να πατάξουμε τη ρήπανση και το, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ήρθε η στιγμή να δράσουμε. Και αν δεν είμαστε έτοιμοι, ειλικρινά, είμαστε απλώς υποκριτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γεωργίου, παρακαλώ. Κυρία Φόντερ Λάιεν, θυμηθήκατε και σήμερα το σιδηρούν παραπέτασμα. Το θέμα μας και το θέμα σας δεν είναι το σιδηρούν παραπέτασμα το θέμα σας είναι η ανεργία και η εξαθλίωση των Ευρωπαίων πολιτών, του ασθενικό κοινωνικό κράτο, η στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, η κλιματική κρίση, η τραπεζική δικτατορία στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Το θέμα σας είναι τα ψεύτικα και θεατρικά λόγια όταν αντιμετωπίζουμε τις αφόρητες προκλήσεις του Ερτογά στην Κύπρο, στη Λιβύη και στη Συρία, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των λαών της περιοχής είναι το αιματηρό μοίρασμα των ενεργειακών πόρων στην περιοχή είναι όταν λέτε και λέμε στον ερντογάν ότι είναι στρατηγικός μας εταίρος όταν του πουλούμε όπλα και όταν διαπραγματευόμαστε το προσφυγικό της ψυχές των ανθρώπων δηλαδή εγκλείοντας τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και αυτό πραγματικά είναι όντως έναν είναι αυτόν ένα, με ακούτε είμαι βέβαιο. έναν σιδηρούν παραπέτασμα που αποτελεί ντροπή και ηθικό πλήγμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να τηρούμε το χρόνο μας, γιατί αυτή τη στιγμή κινδυνεύει και το κατσιάι. Και ξέρω ότι κινδυνεύει και η ζωή μου που σας το ανακοινώνω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Και ζητώ συγγνώμη. Για ένα λεπτό, κύριος Ραντατσόφσκι, παρακαλώ vážení kolegovia osobne som presvedčený είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να αποτύσσουμε φοροτιμήσει στον λαό της Μεγάλης Βρετανίας στον κύριο Φάρατσε και στο κόμμα του Brexit που μας έδειξαν τον δρόμο. Ε, ποιος είναι ο δρόμος ε, στον οποίο θα πρέπει να πάει μια πολιτισμένη και δημοκρατική Ευρώπη. Στο ε, το Ηνωμένο Βασίλειο φέρνει βγει από την Ευρώπη, από τις μη δημοκρατικές θεσμικές διαδικασίες. Είμαι πεπισμένος ότι ότι στο άμεσο μέλλον ε, θα έχουμε μια συνεργασία ε, μεταξύ κρατών, κυρίαρχων και ελεύθερων. Δεν θα έχουμε την ε, μη δημοκρατική διακυβέρνηση από τις Βρυξέλλες πλέον. Ο κύριος Κασπάρη για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μίλησαν για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Ακριβώς αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Θάρρος, ένα προσανατολισμό, ιδέες, ηγεσία. Ευχαριστούμε την κυρία Φοντερ Λάιεν για τις προτάσεις της. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για να πάει μπροστά η Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Συμβούλιο όμως αξιότιμε πρόεδρε του Συμβουλίου κύριε Μισελ, στην τελευταία εκλογική ε, περίοδο και ο κύριος Γιούγκερ είχε εξαιρετικές ιδέες, όμως το πρόβλημα ήταν πόσα μπορέσαμε και πόσα δεν μπορέσανε να κλείσουν από το Συμβούλιο λόγω των αποφάσεών τους. Πόσες ε, καθυστερήσεις υπήρχαν, πόσα μπλοκαρίσματα στο Συμβούλιο, γιατί δεν ε, λάμβανε αποφάσεις. Πόσες ε, χώρες ε, αμφισβητούσαν τα όσα συμβαίναν γιατί υπήρχε πρόβλημα με το πώς ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό για τα ζητήματα της έρευνας, ε, για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό εσπευμένα σας ζητώ να κινητοποιήσετε το Συμβούλιο γιατί αυτή την κινητοποίηση τη χρειαζόμαστε άμεσα και στην Ευρώπη. Η κυρία Ντάλη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2050, για την ουδετερότητα στο κλίμα. Αρνήθηκε να υπογράψει η Πολωνία. Και αυτό δεν είναι ομοφωνία, ακόμα και αν προσπαθεί να το βαφτίσει έτσι το Συμβούλιο. Είναι ζήτημα χρόνου, αλλά ελπίζω όλα τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν. Ελπίζω να φτάσετε σε αυτούς τους στόχους, να έχετε το θάρρος να πιέσετε με φιλόδοξα μέτρα από τώρα και να μην αφήσετε το δίδυμο των μεγάλων κρατών μελών να κυβερνήσουν. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν πιστεύουν όμως τα κράτη-μέλη ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουν, τότε θα πρέπει να βάλουν και το χέρι στην τσέπη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις, αλλά οι προκλήσεις γίνονται ευκαιρίες αν είμαστε ενωμένοι και βρούμε το σωστό δρόμο να προχωρήσουμε. Και τα τρία θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη όλοι μαζί. Ευχαριστώ, κυρία Αγέ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 2.337 δις. Αυτή είναι η τεράστια τρύπα που χωρίζει στον προπολογισμό τα κάτι μελη από το Κοινοβούλιο. Η Φινλανδία δημιούργησε περισσότερους διχασμούς. Δεν ικανοποιήσατε την πλειοψηφία των κατομελών ε, και το κοινοβούλιο που θέλουν περισσότερο, ούτε μια μειονότητα που θέλει λιγότερα. Ε, και τελικά οι νέε φιλοδοξίε τη Επιτροπή ε, δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων και των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πού να βρούμε τα χρήματα. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Μπορείτε λιγάκι να επιβραδύνετε. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ε, Πού θα βρούμε τα χρήματα είναι άλλο από Ευαγγέλιο. Ε, κύριε Μισελ, οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν την ευθύνη ε, να επιλύσουν, σα ανέθεσαν την ευθύνη να επιλύσετε τον τραγωνισμό του κύκλου ως πρόβλημα. Ε, θα περάσετε πολλά άγρυπνα βράδια. Το Κοινοβούλιο θέλει να περάσουμε σε επικοδομητικέ προσπάθειε και να σα βοηθήσει. Διότι τώρα έχετε μια εξίσωση άλυτη να λύσετε. Και εμεί ξέρουμε την απάντηση. Ήδη πόροι. Χρειαζόμαστε οικονομική αυτονομία, δημοσιονομική αυτονομία και θέλουμε πόρου που να συμβάλλουν στην επιτέξη των πολιτικών μα στόχων και να μα επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε το περιθώριο ελληνικού. Εκεί θα συναντηθούν κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, του ίδιου πόρου. Δεν είναι το πρόβλημα οι διπόροι, είναι η υπέρτατη λύση και για αυτό το λόγο δεν θα δώσουμε τη συμφωνία μα εάν δεν υπάρξει πρόοδο σε αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δυστυχώς όλα αυτά που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ότι καλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, και το λαό του. Όμω τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την σκληρή πραγματικότητα του Brexit. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε τη δέσμευσή του να δημιουργήσει ισότιμου κανόνε παιχνιδιού, ε, ξαναβλέποντα του κανόνε εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειου. Όμω η Βρετανική κυβέρνηση ήδη απειλεί να μην τηρήσει τι υποσχέσει τη και τα συμφωνηθέντα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με τα εργασιακά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντο, την κοινοβουλευτική παρακολούθηση των ε, εμπορικών συμφωνιών ε, και την ε, πιθανότητα για ένα Brexit χωρίς συμφωνία τελική στα τέλη του Γενάρη. Το Κοινοβούλιο όμως με τις αποφάσεις του δείχνει ε, τι μπορούν να πετύχουν ε, όλοι οι λαοί, τα έθνη, ε, εργαζόμενα μαζί και κοιτάζοντας να προστατεύσει τους πολίτες από τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών. Διότι η κλιματική καταστροφή, η κοινωνική αδικία και η οικολογική κρίση ακριβώς αυτό είναι που θέλουμε να αναχαιτήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των εκατομμυριούχων και των εταιρικών ομίλων να μην πριτανεύσουν ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να κοιτάξει πώς θα ξεπεράσει και αυτές τις προκλήσεις στο μέλλον μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κύριο κύριος Βιλίμσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Ακούγοντας αυτά που λέτε, έχω την αίσθηση ότι για σας παρά τα αρνητικά επιτόκια και τα μηδενικά δεν έχουμε κρίση νομισματική, κρίση εργασιακή, κρίση οικονομική, κρίση μεταναστευτική. Μία κρίση υπάρχει μόνο, η κλιματική. Ας έχει. Ας το συζητήσουμε αυτό. Αυτό το περιγράψατε την περασμένη φορά στο Στρασβούργο ως έκτακτη ανάγκη. Για μένα αυτό είναι υπερβολές και ιστερίες. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πλειοψηφία γι' αυτό. Ε, η ευρωπαϊκή νομεκλατούρα όμως όταν παίρνει αεροπλάνα και πηγαίνω έρχεται για να συνεχίσει να ε, συζητάει. Είναι δικό σας πρόβλημα. Εκεί που θα μπορούσατε να έχετε αποτέλεσμα είναι αυτή η συζήτηση για την ενιαία έδρα. Να σταματήσει αυτό το πηγενέλα, να εγκατασταθούμε κάπου. Βρυξέλλες ή Στρασβούργο και όχι αυτό το αιώνιο τσίρκο περιφερόμενος θείασος. Κατεβείτε ε, λίγο εδώ στο υπόγειο, στον γκαράζ Κοιτάξτε στον καράζ ε, των βουλευτών. Ε, τι αυτοκίνητα έχουμε, σαν να γυρνάμε την ταινία Fast and Furious στο επόμενο επεισόδιο και όχι προστασία. Ε, κοιτάξτε τι αυτοκίνητα έχουμε. Ο κύριος Έπινγκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μισελ, γνωριζόμαστε. Είστε απογοητευμένος για ε, τη Μαδρίτη και τη Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα. Μα είναι 27.000 ε, οι ε, σύνεδροι εκεί. Πώς να διαπραγματευτείς και ποιο είναι το αποτύπωμα. 60.000 τόνοι διοξίδιο του άνθρακα ήταν αυτή η σύνοδος και λέει ο Guardian και του χρόνου είναι στη Γλασκόβη και αυτή είναι ε, τσίρκο και μετά στο Βανκούβερ, Ντέρμαν, Καλή, Καζάν, Έντιμπορ, Κιώτο και πάει λέγοντας. Αυτό κύριε και κύριοι φαίνεται ε, να είναι Φόρμουλα 1, ε, όχι σύνοδος για το κλίμα και και μπορώ να σας πω ότι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα το, της Φόρμουλα 1 εκπέμπει λιγότερο. Το 2030 θα είναι κλιματικά ουδέτερο. Ε, Σταματήστε λοιπόν ε, να κάνετε αυτές τις ακριβές διασκέψεις. Εκατό εκατομμύρια κοστίζει κάθε σύνοδος κορυφής για το κλίμα. Ε, προσαρμοστείτε στις εκπομπές της Φόρμουλα 1 επιτέλους. Ευχαριστώ για ένα, για ένα, για ένα λεπτό κύριος ε, Φαράς. Μετά από 3,5 χρόνια δράνειας ε, και καθυστερήσεων θα φύγουμε από αυτή τη φυλακή των εθνών στα τέλη του Ιανουαρίου. Δεν θα γίνουμε τρίτη χώρα, όπως είπατε. Όχι, θα είμαστε μια ανεξάρτητη, αυτοδιατηθέμενη και αυτοκυρίαρχη χώρα. Ε, νομίζω ότι αυτά τα ξέρετε πολύ καλά, αλλά συνήθως ε, ε, δεν το λέτε. Γενικά δεν θέλουμε να έχουμε πρόσωπους ε, γραφειοκράτες που μας κυβερνούν. Το ακούσατε, σας απορρίπτουν. Είναι πολύ τα νέα συγκεκριμένα έχουμε ε, αυτή την πλειοψηφία στις εκλογές η οποία μας βγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit θα είναι η αρχή του τέλους αυτού του εγχειρήματος. Τώρα η Ευρώπη των κυρίαρχων κρατών θα πρέπει να συνεργαστεί, να είναι φίλοι, τους, φίλοι μεταξύ τους, αλλά να μην ε, κάνουν τίποτε άλλο. Um, Δεν είναι πολύ ωραίος τρόπος για να βρείτε καινούριου ε, φίλους αν μιλάτε για Ότι, ότι οι συνάδελφοι που μιλάνε για τα θέματα αυτά είναι βαρετοί σαν ε, του θανατά. Ε, εδώ λοιπόν, όπως ε, όλοι εδώ έχουμε πρόσωπα και αυτοί που εσείς είπατε αόρατους ή ασήμαντους είναι εκεί έξω και αγωνίζονται για τον Brexit. Εγώ λοιπόν πρέπει να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και του θεσμικού μας οργάνου. κύριε Όλμπριχτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώς να πω ότι είμαι από την Πολωνία και πραγματικά ευνηδιάζομαι από αυτό που μόλις άκουσα. Ποιο, ε, δημοψήφι, ποιο, ποια δημοσκόπηση στην Πολωνία, ποιοι θέλουν να φύγουν από την Ευρώπη. Καινούριο μου φαίνεται, για άλλη χώρα θα μιλάτε. Επίσης, να συνεχίσω στα πολωνικά. Ε, κύριε Πρόεδρε, τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μου ευγνωμοσύνη για τον πρόεδρο γιατί είπατε και χθε ότι θα δεσμευτείτε να συζητήσετε και με εμά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχετε δεσμευτεί για τη μελλοντική μα συνεργασία. Έπειτα, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προ το Συμβούλιο για το γεγονό ότι δεν μας έκλεισε την πόρτα στα μούτρα μετά την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας. Διότι πραγματικά αυτό ήταν απλώς ένα σημείο αφετηρίας, αλλά δεν είναι καλή βάση για τις μελλοντικέ μας συζητήσεις. Καλό θα ήταν λοιπόν το Συμβούλιο να μην πετάξει όσοι έχουν γίνει ως τώρα, αλλά αυτή την πρόταση να τη θάψει για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και μετά για το Brexit, μια σοβαρή πολιτική απόφαση που έχει να κάνει και με τα μελλοντικά του προπολογισμού και τα δημοσιονομικά. Ευχαριστούμε ο κύριος Σίλβα Περέιρα εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών καθίσταται σαφέ ότι στη Βουλή των Κοινοτήτων υπάρχει επαρκή πλειοψηφία για να εγκριθεί η Συμφωνία Αποχώρηση και ε, το Brexit να ολοκληρωθεί ως το τέλος Ιανουαρίου. Βεβαίω είναι μια στιγμή ε, θλιβερή για το μέλλον της Ευρώπη, αλλά είναι και μια δημοκρατική επιλογή που πρέπει να τη σεβαστούμε. Και βεβαίω ε, ο κύριο Φάραντ κάνει λάθο όταν λέει ότι η Ευρώπη είναι μια φυλακή των εθνών. Καθήκον μας τώρα είναι να συγκεντρωθούμε ε, στο κοινό μας μέλλον. Και αυτό σημαίνει να διαπραγματευτούμε με το Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο φιλικό για μια εύρωστη και που να μπορεί να λειτουργήσει με εμπορική σχέση και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της ε, νέας αγοράς και τα υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής, ε, κοινωνικής και εργασιακής προστασίας. Αυτά είναι σημεία κλειδιά για τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις και μόνο μέχρι το τέλος του 2020 θα γνωρίζουμε εάν ε, έχει πραγματοποιηθεί το σενάριο της αποχώρησης χωρίς συμφωνία το no deal Brexit. Τώρα για να επικεντρωθούμε στο κοινό μας μέλλον. Πρέπει να σκεφτούμε τις προσδοκίες των πολιτών μας, να σκεφτούμε σοβαρά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί είναι σημαντικές προτεραιότητες, αλλά υπάρχουν ε, καθυστερήσεις ως προς τις διαπραγματεύσεις του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του Brexit. Με συγχωρείτε, απλώς να πω ότι έχουμε τουλάχιστον 17 ε, συμμετέχοντες στη δικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Δεν λέω ότι δεν θέλω άλλους αγορητές, απλώς να πω ότι πραγματικά γινόμαστε πάρα πολύ ε, αυτοί που λέτε ότι θέλετε να μιλήσετε. Κυρία Λατίνγκα. Ναι, Νέτσιγκα για ένα λεπτό. Όπως είπαν πολλοί, υπάρχει τραγική σαφήνεια για το Brexit. Ε, όμως ε, δεν είναι μόνο ο Μπόρις που πήρε την πλειοψηφία. Υπάρχουν και πάρα πολλοί που ψήφισαν για τα υπόλοιπα ε, κόμματα που ήταν κατά του Brexit. Το, το σύστημα του έδωσε την πλειοψηφία και θα φύγουμε 31η Ιανουαρίου. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Παρνιέ και σε όλους ε, όσους ε, προσπάθησαν να κρατήσουμε στενή τη σχέση μας. Ε, ειδικά με ε, λυπεί ο αντίκτυπος στην έρευνα, στον ακαδημαϊκό χώρο. Μπορέσαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε την επιστημονική τεχνολογική γνώση προς όφελος όλου του κόσμου. Ξέρω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θεωρούν ότι θα προσπαθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο να υποσκάψει τα στάνταρτ για το περιβάλλον και την ε, προστασία των εργαζομένων. Θα προσπαθήσουμε εμείς να διατηρήσουμε όλα αυτά στο Κοινοβούλιο, όπως και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, σας ευχαριστώ όλους που υποστηρίξατε εμάς που παλέψαμε για να μείνουμε πιστεύαμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε καλύτερο μέλλον εντός της Ένωσης. Έχει κάνει λάθος ο κύριος ε, Φαράτς. Η Ένωση είναι ένας φανταστικός θεσμός και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα επιστρέψουμε εδώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Άντερσεν. Ευχαριστώ. Για την ε, ουδετερότητα ε, του κλίματος το 2020 όλοι συμφωνούν. Ο κύριος ε, Λουί Μισελ πράγματα που με χαροποίησαν. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι κάτι που θα μας φέρει προς το μέλλον. Πόσα όμως από αυτά φαίνονται μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν έχουμε τα σωστά κονδύλια για το μέλλον της Υπήρου μας η πρόταση λοιπόν για το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ ε, πολύ μικρή, πολύ λιτή, 25% για την προστασία του κλίματος, ε, για την ψηφιοποίηση. Πώς θα προχωρήσουμε. Μία γεωργία που θα είναι ουδέτερη σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής, ε, τα κτίρια, οι συνδέσεις, οι ε, μεταφορικές συνθέσεις, όλα αυτά ε, πρέπει να έχουν χώρο στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κυρία Φοντερ Λέιεν, παρακαλώ αφήστε μας να διαμορφώσουμε μαζί μαζί ε, όλους αυτούς τους στόχους και στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε κυρία Πιτσότο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρώπη σα είναι πάντοτε υποδουλωμένη στι τράπεζε και τα συμφέροντα τη Γαλλία και τη Γερμανία. Στο τελευταίο συμβούλιο φάνηκε αυτό από τη στάση των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων. Η Γερμανία θέλει μια Ευρώπη με, που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τη. Δεν υπάρχει αυτό που περιγράφεται με τη βράσινη Συμφωνία. Είναι μια μεγάλη μπλόφα και θέλετε ουσιαστικά και ε, με την συνενοχή της δικής μας κυβέρνησης, ε, των σοσιαλιστών και των πέντε αστέρων, να εκμεταλλευτείτε και τους Ιταλούς. Δηλαδή τα συμφέροντα της Ευρώπης να πετανεύσουν σε σχέση με τα συμφέροντα των Ιταλών. Με ε, τις νέες αποφάσεις το 2011 έχετε βάλει το χέρι στην τσέπη των Ιταλών φορολογουμένων. Όμως ε, ποιοι θα προστατεύσουν τους πολίτες, οι γραφειοκράτες των Βρυξελών. Πρέπει εσείς να ετοιμάσετε τα μπαγκάζια σας γιατί πολύ γρήγορα τώρα άμεσα ο Ιταλικός λαός θα σας στείλει σπίτι σας για πάντα. Ένα λεπτό για τον κύριο Βαν Οβερτφέλτ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, η φιλοσοφία πίσω από το Green Deal ε, χρήζει στήριξη, γιατί χρειαζόμαστε ένα, μια βιώσιμη, ρεαλιστική μετάβαση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική πρόκληση. Και το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του σωστά αναφέρει ότι είναι απαραίτητη η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία. Όπω είπε και η Επίτροπο Βερστάγκερ αυτήν την εβδομάδα πολύ σωστά, η τεχνολογία δεν είναι ένα εκτραδάκι για να μα βοηθήσει να προσεγγίσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική ε, αλλαγή. Είναι απαραίτητη. Όμω όλα αυτά συνάδουν και με την ε, χρηματοδότηση και εδώ υπάρχουν ε, διάφοροι άγνωστοι παράγοντε. Σίγουρα και με το ΠΔΠ χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα πάνω από τα 360 δις που αναφέρονται αυτή τη στιγμή. Επομένω, περιμένουμε τα μέτρα χρηματοδότηση. Για το πολιτέ νοσοκομικό πλαίσιο, ο πρόεδρο ε, Μισελ είπε ότι σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή θα πρέπει να βρούμε συμβαστική λύση. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Προέδρου στο γεγονό ότι και το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί στην προσπάθεια εξέβριση αυτού του συμβασμού. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μοντή, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μάλλον είναι η τελευταία μου ομιλία στο Κοινοβούλιο και θέλω να πω ότι εγώ είμαι Σκοτσέζος, είμαι Βρετανός και εγώ παραμένω Ευρωπαίος. Μπορεί να κάθεστε εκεί και να αμφισβητείτε τα όσα λέω. Αλλά εγώ εδώ και πολλά χρόνια υποστήριξα ε, και τα μέλη του Σολινταρνόσκα ε, τη δεκαετία του Όμω εδώ δεν είμαστε σωστοί Ευρωπαίοι σε αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιβαίνει στα συμφέροντα των ε, εργαζομένων και των οικονομιών. Δεν έχει καν να κάνει με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης. Όλο ένα και άοκ να εργάζεται για να ομογενοποιήσει τους πάντες σε ένα κέντρο ε, ολικού ελέγχου. Εμείς Φεύγουμε λοιπόν όχι εξαιτία του Ντόμινι Κάμινγκ ή άλλων, αλλά επειδή ο Νάτζελ Φάρατ και άλλοι δημιούργησαν το κόμμα του Brexit και πέτυχαν το Brexit. Κόβεται το μικρόφωνο. Ο κύριος Μπόκταν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια στιγμή παρακαλώ. Με συγχωρείτε Παρακαλώ, συνάδελφοι. Καταλαβαίνω τι ότι με την ελευθερία καθώ είμαι Ιρλανδή. Ο κύριος Μπογκδάν. Η Ρωμανία ε, αποφύγει το μαθηματικό κριτήριο που ακολουθεί η Φιλανδική Προεδρία για τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε ότι ε, το σχέδιο του προπολογισμού εκφράζει ένα όραμα το να μιλάμε για περικοπέ χωρί να λαμβάνουμε υπόψη τι ανάγκε των κρατών μελών. Ε, σημαίνει ότι μεγαλώνουμε το χάσμα μεταξύ Ανατολή και Δύση και υποσκάπτουμε την έννοια τη συνοχή. Η αρχή μεταφορών κονδυλίων μεταξύ των ταμείων αυξάνει τη γραφειοκρατία Γι' αυτό η σημερινή πρόταση για τη συνοχή και για την κοινή αγροτική πολιτική δεν μπορεί να υποστηριχθεί από τα κράτη τη Ανατολική Ευρώπη. Η Ρουμανία δεν υποστηρίζει την Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Έχει μία ταχύτητα η Ευρώπη. Υποστηρίζουμε την ιδέα της επίτευξης κλιματικής αλλαγής ε, μέχρι το 2050. Μιλάμε για ένα φιλόδοξο αλλά πολύπλοκο στόχο ταυτόχρονα και απαιτούνται κατάλληλα μέτρα ε, για το κάθε κράτος μέλος. Υπάρχουν ε, πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των πολιτών ανάλογα με το κράτος μέλος. Σας ευχαριστώ. κυρία Φρίτσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει το στόχο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Πράγματι απαιτείται δράση από μέρους μας και μάλιστα άμεση δράση. Οι χώρες ε, παγκοσμίω ε, δεν μπόρεσαν να έρθουν σε μια συμφωνία και πολύ απογοητευτήκαμε και Γι' αυτό είναι όλο ένα και πιο σημαντικό για μα να έχουμε ένα κοινό στόχο. Θέλουμε να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση κλιματικά ουδέτερη. Αυτό είναι ο στόχο μα. Και αυτό συνάδει με τη Συμφωνία του Παρισιού. Σημαίνει μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει νέε ευκαιρίε, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέε αγορέ, νέε τεχνολογίε. Και φυσικά νέε ευκαιρίε και επιπρόσθετα μια νέα πράσινη ανάπτυξη για μας. Εδώ ε, έχει έρθει και θα μείνει η πράσινη μετάβαση. Θα πρέπει να είναι ευφυής και δίκαιη και θέλω να διασφαλίσω ότι όλοι εμείς θα πιέσουμε γι' αυτό. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πρώτη η Ήπειρος που θα είναι κλιματικά ουδέτερη. Ευχαριστώ κυρία Χρεαντζόβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από την αποτυχία της COP25 στη Μαδρίτη, η Ευρώπη φαίνεται να είναι μία από τις ε, ε, λίγες χώρες, λέει μιλήτρια, που θέλει να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή. Αυτό Όμω θα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να ενθαρρύνουμε και άλλου εκτό τη Ευρώπη ε, να κάνουν αυτό που του αναλογεί. Η Κίνα, λόγου χάρη, δεν μπορεί να ορίζεται πλέον ω αναπτυσσόμενη χώρα. Η Ευρώπη δεν θα σώσει μόνη τη τον πλανήτη. Η τσεχική δημοκρατία θέλει να συνεισφέρει για το κλίμα, αλλά θα χρειαστούμε βοήθεια. Η πρόταση για το Ταμείο Μετάβαση δεν θα πρέπει να αφορά το Ταμείο Συνοχή με μια νέα ετικέτα. Θα πρέπει να μιλάμε για νέα ταμεία. Επίση, καλή ιδέα είναι το Πράσινο Ταμείο Ανάπτυξη, αλλά χωρί τον ιδιωτικό τομέα δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τι ανάγκε των βιομηχανοποιημένων χωρών, όπω είναι η Σλοβακία, η Τσεκία και άλλε χώρε τη περιοχή που αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερη πρόκληση για να πετύχουν τους κλιματικούς στόχους, ενώ θα διατηρήσουν και την οικονομική τους ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κυρία Φίλιπς, για ένα λεπτό. Well, I see the European Parliament has already βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει να περικόπτει τις εκπομπές ε, Υποτίθεται ότι το πιστεύετε αυτό, αλλά αυτό είναι αστείο. Για τρία ολόκληρα χρόνια ήσασταν ε, τελείω παράλογοι. Ασκήσατε εκφοβισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Βρετανοί δεν θα αλλάξουν γνώμη. Έτσι, να το ξέρετε αυτό, γιατί κάνατε απόλυτα λάθο. Οι ψηφοφόροι δεν ζουν μέσα στη δική σα τη φούσκα. Δεν θέλουν ψέματα. Ε, δεν θέλουν φανατικού. Και παρά τι προσπάθειέ σα, το Brexit θα στεφτεί από τεράστια επιτυχία επιτυχία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βάρο στις διαπραγματεύσεις και ελπίζω ο Μπόρι Τζόνσον θα σα δείξει ότι πρέπει να ξεχάσετε του ίσους όρου ανταγωνισμού. Εμεί θέλουμε ελευθερία. Εμεί δεν είναι απλά ότι θα επιβιώσουμε, αλλά θα ευημερίσουμε. Αντί να αποφεύγει το αντίνατο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο που θα είναι πραγματικά δημοκρατικό και παγκοσμιοποιημένο και να μην το ξεχνάτε. Οι φεντραλιστέ θα δουν το δικό σα το ηλίθιο εγχείρημά σα να εξαφανίζεται. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλό Brexit. Η κυρία Τότε για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν, συμφώνησαν στο πνεύμα της κλιματικής ουδετερότητας το γεγονός ότι η Ευρώπη μέχρι το 2015 θα είναι ουδέτερη ως προς το θέμα του κλίματος. Αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν και πρέπει να, να ορίσουμε τις βασικότερες προδιαγραφές. Ένα όρος είναι ότι δεν θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι αλλά οι επιχειρήσεις και τα κράτη που αυτά κατ' ουσίαν μολύνουν, τη, ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Το κόστο, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τι οικογένειε. Είναι οι κανόνε δεν θα πρέπει να οδηγήσουν στο να αυξηθεί το κόστο για τα τρόφιμα. Άρα δηλαδή τα φτωχότερα κράτη δεν θα πρέπει να λάβουν λιγότερα κονδύλια από το Ταμείο συνοχή, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο απλά θα επιταθεί η ανισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να επιδιώξουμε να μειωθούν οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μια ουδέτερη τεχνολογία. Και τέλος θέλω να επισημάνω ότι η Ουγγαρία ε, αποδεικνύει όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις ότι επιθυμεί να είναι ουδέτερη ως προς το κλίμα. Διότι τις εκπομπές μας του διοξιδίου τις μειώσαμε κατά 30%. Μάρκες, για ένα λεπτό. Να πω εδώ κάποια σύντομα λόγια για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς ε, πρέπει να δούμε πόσο χρόνο αφιέρωσαν οι ηγέτες αυτή τη συνεδρίαση για το ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ. Αυτό το Συμβούλιο ήταν μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους ηγέτες να φτάσουν σε συμφωνία για ένα προπολογισμό που είναι θεμελιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μένει στα χέρια του Πρόεδρου Σαρλ Μισελ να κάνει αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη εδώ η χθεσινή μα συνεδρίαση και η δική του πρωτοβουλία με τον πρόεδρο όλοι ήταν ένα πρώτο βήμα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί από τον Νοέμβριο πέρσι και η συνένεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο απαιτεί πολιτική συμφωνία για τους ίδιους πόρους για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ε, Πρόεδρε, η πρόταση του Συμβουλίου που είναι επιτάπητος είναι παράδεκτη. Θέλουμε ένα προϋπολογισμό τον Ιανουάριο του 2020, αλλά δεν θα είμαστε σε θέση να συμβιβαστούμε με, αυτό τον, ε, με αυτή την πρόταση. Ο κύριος Κέλεχερ για ένα λεπτό. Οι βρετανικέ εκλογέ ε, ήταν ε, μια ξεκάθαρη και αποφασιστική νίκη για το κόμμα των συντηρητικών. Το Μήνο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα περάσει η Συμφωνία αποχώρηση και θα φύγουμε στις 31 Ιανουαρίου. Υπάρχουν και ρήτρε προστασία ε, για να μην υπάρξει ξεκάθαρο σύνορο ε, με την Ιρλανδία και αυτό είναι πολύ καλό. Όμω ο κύριο Μπανιέ θα πρέπει να μην εφησυχάζει, να διασφαλίσει ότι οι συζητήσει θα συνεχιστούν και μετά την συμφωνία αποχώρηση για να μην υπάρξει σύνορο στο νησί. Ε, πρέπει να διατηρηθεί και η συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή γιατί οι πολίτες εκτιμούν ιδιαίτερα και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Να έχετε κατά νου ότι πολλοί Βόρειοι Ιρλανδοί θέλουν να εξεκαθαρίσουν και να ε, εκφράσουν την ταυτότητά τους και ω Ευρωπαίοι πολίτες. Η πλειοψηφία των πολιτών μα το θέλει αυτό. Υπάρχει μια νέα ευθυγράμμιση στην Βόρεια Ιρλανδία ε, και σίγουρα αλλάζουν και τα δημογραφικά στοιχεία και θα έχουμε ε, νέου πολιτικού συσχετισμού ε, στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν να δικαιωθεί η Συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή και να προωθηθούν προτάσει που θα διασφαλίσουν ένα δημοκρατικό μέλλον για την Βόρεια Ιρλανδία. Ο κύριος Μημεράκης, για ένα λεπτό καλωσορίζω τα συμπεράσματα του συμβουλίου σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την παράνομη συμφωνία μεταξύ τουρκίας και λιβύης διότι η στήριξη που έλαβε η ελλάδα και η κύπρος από την ευρωπαϊκή ένωση αποτελεί ένα βήμα σημαντικό για τη σταθερότητα της μεσογείου αλλά και για τη θωράκιση των θαλασσίων συνόρων μας. αποτελεί επίσης ισχυρή απόδειξη με επιχειρήματα και απάντηση στους αβάσιμους ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς. παρά τα αυτά όπως έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν η τουρκική κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου στη συγκεκριμένη περίπτωση το δίκαιο της θάλασσας και συνεχίζει επιθετικά μια πολιτική στρατηγική η οποία καταπατά κάθε κανόνα και κάθε κεκτημένο. και με τις προκλητικές τους αυτές παρεμβάσεις η τουρκία και ο πρόεδρος ερντογάν αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της μεσογείου και κατ' επέκταση της ιδείας της ευρώπης. συνεπώς η συμπεριφορά του περιφερειακού ταραξία πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιαία συντονισμένα άμεσα και με κυρώσεις. είναι ανάγκη να εξετάσουμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεών μας με την τουρκία και να αποδείξουμε έμπρακτα ότι η ευρώπη δεν είναι απλώς θεατής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον πρόεδρο Μισελ όταν μίλησε για την συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και είδα και τα συμπεράσματα. Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέχρι πρόσφατα ε, δεν είχε φιλοδοξίες και κύριε Μισελ είχα την ελπίδα ότι και εσείς θα συμβάλλετε έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η στάση του Συμβουλίου κατά το επόμενο έτος. Γιατί αυτή η διάσκεψη είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία ε, να σταθεροποιηθεί η Ευρώπη και εφόσον μας εγκατέλειψαν αυτοί που είναι υπέρ του Brexit να έχουμε επιτέλους μια νέα αρχή στην Ευρώπη. Όμως για να το επιτύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα θαραλέο φιλόδοξο σχέδιο και οφείλουμε πράγματι να ε, συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες. Δεν αρκεί λοιπόν να παραπέμπει κανείς στην στρατηγική ατζέντα ούτε ε, να περιορίζεται στο να λέει τι έχει πετύχει μέχρι τώρα. Εγώ θα ήθελα να πω αυτό που είχε πει κάποτε ο Βίλι Μπραντ, να υπάρχει περισσότερη δημοκρατία με νέα αρχή σε αυτό το θέμα κατά το νέο έτο και στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, καταθέσουμε ένα καλό φιλόδοξο σχέδιο έτσι ώστε να διεκδικήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ κύριο για ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να εκφράσω την χαρά μου που βλέπω ότι η Κομισιόν υιοθετεί την ιδέα της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας συνδέοντας την Πορτογαλία με την και την Ισπανία με την υπόλοιπη Ευρώπη στα σύνορα των Πυρηναίων και το θέτει αυτό ως προτεραιότητα για τον Green Deal. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο οικολογικό, οικονομικό ζήτημα, αλλά είναι και γεωπολιτικό. Εμείς θα εξαρτώμαστε λιγότερο από τη Ρωσία αν ανοίξουμε τις πόρτες της ε, Ευρωπαϊκής Ενέργειας στην Ιβρική Χερσόνησο, γιατί πρόκειται για καθαρή ενέργεια που μπορεί να εισαχθεί από άλλε περιοχέ και θα μειώσουμε την εξάρτησή μα από τη Ρωσία. Θέλω να χαιρετήσω και τον πρόεδρο Σελμίσερ και να πω ότι είμαι κάπω απογοητευμένο από την έλλειψη οράματο ε, του Συμβουλίου σε σχέση με το μέλλον τη Ευρώπη. Είναι σημαντικό ε, το Συμβούλιο εδώ να παίξει ρόλο και θα πρέπει και το Κοινοβούλιο ε, να ακουστεί. Πρέπει να ακούσουμε πρώτα τους ε, πολίτες. Ε, δεν πρέπει να παρουσιάσουμε αποτελέσματα πριν να ακούσουμε τους πολίτες. Γιατί λοιπόν εμείς είμαστε καλή την πίστη να συνεισφέρουμε, αν το Συμβούλιο το επιθυμεί βεβαίω. Ευχαριστώ κύριος Μαυρίδης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα συμπεράσματα υπήρξε ομόφωνη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιβεβαίωσε την παράνομη συμπεριφορά της τουρκίας τόσο στην κυπριακή αος όσο και με το λεγόμενο μνημόνιο με το καθεστώς της τρίπολης και στις δύο περιπτώσεις η τουρκία ενεργεί έξω από το διεθνές δίκαιο και έξω από το δίκαιο της θάλασσας του οηε. σήμερα όμως το συμβούλιο επανέλαβε την αλληλεγγύη του προς τα κράτη μέλη των οποίων τα κυριαρχικά δικαιώματα παραβιάζονται επί της ουσίας η επίθεση του Ερτογάν είναι ενάντια στην ευρωπαϊκή ένωση είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο το οποίο αποτελεί κοινοτικό κεκτημένο και πλήττει τα ύψιστα στρατηγικά συμφέροντα της ευρωπαϊκής ένωσης τα οποία περιλαμβάνουν σχεδιασμούς για την ενέργεια στην ανατολική μεσόγειο. ωστόσο όμως καθώς σήμερα μιλάμε αυτά τα θέματα το συμβούλιο και καθώς το συμβούλιο αποφάσισε μέτρα κατά της τουρκίας αύριο η νέα επιτροπή ξεκινά διάλογο για αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων με την τουρκία. ο Ερτογάν θα δημιουργήσει νέο τζιχαντιστικό καθεστώς στη λιβύη και εμείς πρέπει να προασπιστούμε τα ύψιστα συμφέροντά μας. Συνάδελφοι, πρέπει να πω ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κατσδιά, γιατί πρέπει να περάσουμε αμέσως στην απονομή του βραβείου Ζαχάρου στις 12 το μεσημέρι και λυπάμαι για όσους ήθελαν να μιλήσουν. Η κυρία Νίμπλερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμη Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω δύο παρατηρήσεις για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είπαν τίποτα για την κατάσταση στη Μάλτα. Και μιλάμε εδώ για πληρωμένη δολοφονία στη Μάλτα, όπου έχουν εμπλακεί και κυβερνητικά στελέχη. Εγώ το λέω ξεκάθαρα όνειδος και ντροπή. Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Η Πράσινη Συμφωνία ε, θέλουμε να είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες, σε ευφύς ε, λύσεις και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε μέχρι το 2050 να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Τεχνολογικά αυτό είναι δυνατόν, όμως όλα αυτά θα πρέπει να έχουν και οικονομικά νόημα φοβάμαι ότι η πολιτική του κλίματο και η πολιτική για τον ανταγωνισμό είναι δύο διαφορετικά πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που παράλληλα με την πρόταση για το κλίμα θα παρουσιάσετε και τη βιομηχανική σα πολιτική. Αυτό είναι μια καλή δήλωση και με μεγάλη περιέργεια περιμένω να ακούσω τι προτάσει σα. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ο κύριο Κόρμπετ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καθώς προχωράει η διαδικασία του Brexit, παρακαλώ να έχετε κατά νου και να θυμάστε ότι το 53% ψήφιζε σε αυτές τις εκλογές. Ε, ε, ψήφισε λοιπόν κόμματα που ήθελαν και δεύτερο δημοψήφισμα. Όλε οι δημοσκοπήσει την τελευταία χρονιά, εκτό από μία, έδειξαν ότι η πλειοψηφία των Βρετανών θα ήθελαν να παραμείνουν. Θα είχαν ψηφίσει το Remain αν υπήρχε δεύτερο δημοψήφισμα. Και ο κύριο Τζόνσον, 43% των ε, ψήφων, μόλι 1% παραπάνω από την κυρία Μέη, θεωρεί ότι αυτό είναι λευκή επιταγή για να προχωρήσει σε, ε, σε μια άτακτη αποχώρηση, hard Brexit. Και αυτό θα κάνει, γιατί ήδη έχει πάρει πίσω τη δέσμευσή του ότι η Βουλή των Κοινοτήτων θα ψηφίσει για την παράταση τη ε, μεταβατική περίοδου για να δώσει χρόνο για διαπραγματεύσει. Ήδη λέει ότι δεν θα πάρουμε παράταση. Θα το καταστήσουμε παράνομο δεν θέλει να διαπραγματευτεί λοιπόν μία ε, σωστή συμφωνία εταιρική σχέση. Η στρατηγική του διαπραγματεύσει είναι δώστε μου αυτό που θέλε, θέλω, αλλιώ θα αυτοπυροβοληθώ στο κεφάλι. Τέλο, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον ε, κύριο Βερχόφστατ ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να υιοθετήσει οποια, οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι τη στιγμή που θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα και από τι δύο πλευρέ των πολιτών πάντα. The ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερω που είχατε δυνατότητα να μιλήσω ε, στην ε, συνάντηση του Συμβουλίου το Σαββατοκύριακο και να συμμετάσχω στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την... Χθες το βράδυ ο εξαίρετος ε, Μισελ Μπαγνιέ μα έδωσε, μας διαγράφησε τον επόμενο χρόνο, το επόμενο μήνο και τόσο θα συμβούν. Πρέπει να υπάρχει όμως ε, ε, καλή βούληση και εμπιστοσύνη. Ιδάλω θα αποτύχουν οι πραγματεύσει. Δεν πρέπει λοιπόν να βάζει αυθαίρετα όρια χρονικά ο κύριος Τζόνσον. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει μια σωστή συμφωνία πιο σημαντικό από το να γίνει το Brexit. Ελπίζω να συμβεί αυτό. Ε, συμφωνώ και μετά όσα είπε η Πρόεδρο για το πολιτέ νομικό πλαίσιο. Πρέπει όλοι να ε, σταθούν στο ύψο των περιστάσεων, να έχουμε τον κατάλληλο προπολογισμό. Αλλιώ πρέπει να βρούμε ίδιου πόρου. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών και τώρα θα δώσουμε το λόγο στο Μίσελ Μπερνιέ, ο οποίο είναι επικεφαλή για τι διαπραγματεύσει για τον Brexit. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. το αίτημα της κυρίας Φόντερ Λάιεν, όπως ε, πολύ και εσείς αναφέρετε, ε, με το Brexit και θα ήθελα να δώσω κάποιες ε, απαντήσεις για το θέμα αυτό. Καταρχήν, όπως πολύ είπατε, να παρατηρήσω ότι είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο συζητά το Brexit. Γνωρίζετε ότι πράγματι θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου και το λέω αυτό με πολύ σεβασμό και κατανόηση. Άκουσα και τις παρεμβάσεις των κυρίων Τσόλος, Πέρες, σκατιέλερ. Ε, Πολλοί από εσά εδώ, εκτός του Κοινοβουλίου, θα θέλατε το Ηνωμένο Βασίλειο, θα επιθυμούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως εκφράζουμε και σεβασμό απέναντι στην Βρετανική επιλογή από την αρχή και ε, η ευθύνη μας, η δική μας αποστολή, αυτή η αποστολή που ανέλαβα εγώ, είναι ακριβώς να σεβαστούμε την βούληση που εκφράζεται από την πλειοψηφία των Βρετανών πολιτών και επομένως να οργανώσουμε την τακτική αποχώρηση προς ε, το συμφέρον των πολιτών, της οικονομίας ε, και των δύο πλευρών και προς το συμφέρον του μέλλοντος ε, μέσω μιας συμφωνίας, μιας που βρίσκεται εδώ, τη γνωρίζετε καλά, γιατί ουσιαστικά την οικοδομήσαμε μαζί κατά κάποιο τρόπο. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον Brexit, Brexit Steering Group και όλους τους βουλευτές και κυρίως τον κύριο Φερχόφστατ. Τώρα, ε, είμαστε στραμμένοι προς το μέλλον ε, και η κυρία Φαντελάιεν ε, είπε εδώ στις 27 Νοεμβρίου όποιο και είναι το μέλλον μας οι δεσμοί και η φιλία μεταξύ των λαών μας θα μείνουν ως έχουν αυτό θα μας καθοδηγήσει με ένα τρόπο σεβασμού και με ένα φιλόδοξο τρόπο στο να οικοδομήσουμε ισχυρή στρατηγική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα βασιζόμαστε σε έναν οικονομικό πυλώνα και με τον Φιλ Χόγκαν και με τους ε, άλλους αρμόδιους επιτρόπους. Ε, θα εργαστούμε για το θέμα αυτό ε, και επίσης θα εργαστούμε κατά προτεραιότητα με το Ζωζέ Μπορέλ και τους άλλους επιτρόπους για το στρατηγικό όραμα. Θα μείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμμαχος και φίλος και τέρος, το Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον θα μείνει σύμμαχος και φίλος και θέλουμε να τα εγγράψουμε αυτά σε νέες συνθήκες και συμφωνίες. Το μέλλον αυτής της φιλόδοξης σχέσης έχει καταγραφεί με πολύ ακριβό τρόπο στις 36 τελευταίες σελίδες αυτού του εγγράφου που έχετε ενωπιών σας. Να υπενθυμίσω ότι αυτή ε, η πολιτική, δήλωση είναι κοινή. Κάθε λέξη μετράει και έχει συμφωνηθεί από εμά και από τον Μπόρις Τζόνσον. Κάθε λέξη μετράει, όπως σας είπα. Τι μπορεί να περιορίσει αυτή τη φιλοδοξία, κύριοι βουλευτέ, Δύο πράγματα. Ένα, ο χρόνος. Χρειαζόμαστε χρόνο για να ε, μεταφράσουμε σε κείμενα τις φιλοδοξίες αυτές ε, και δεύτερον οι αποκλήσεις που μπορεί να προκύψουν ε, σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά μας και τους στόχους μας. Πιο συγκεκριμένα τώρα ε, η απάντηση που θα δώσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ερώτηση. Αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόμαστε την επιλογή του, αλλά δεν εγκαταλείπει την Ευρώπη. Θέλει να απομακρυνθεί και σε ποιο βαθμό από το κανονιστικό μας μοντέλο. Και αυτή η ερώτηση τίθεται και θα καθορίσει το πέντε τη φιλοδοξία μα η απάντηση που θα δοθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα έχουμε ε, τρία επίπεδα στα οποία πρέπει να εργαστούμε. Ένα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία τη κύρωση τη συμφωνία αποχώρηση. Δεύτερον, ε, η υλοποίηση τη ίδια τη συμφωνία ε, σε όλε τι διαστάσει. Αυτό δεν είναι αμεληταίο. Ε, ούτε για του πολίτε. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του που εγγράφονται στο κείμενο αυτό και να επενθυμίσω, κυρία Πρόεδρε, το είπα και στον κύριο Κέλλελερ και στον κύριο Κέλλη και σε άλλους στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ερλανδία. Ε, πρέπει να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ειρήνη. Και το τρίτο, τρίτος πυλώνας είναι οι διαπραγματεύσεις στο μέλλον οι διαπραγματεύσει θα λάβουν χώρα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι δεν θα ζητήσει παράταση τη μεταβατική περίοδου. Είναι δυνατή η παράταση αυτή και θα παραμείνει δυνατή μέχρι τι 30 Ιουνίου σε μια κοινή συμφωνία. Δηλαδή, ο κάθε εταίρο, η Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να πούν ναι ή όχι μέχρι τι 30 Ιουνίου. Όμω είναι περιορισμένο ο χρόνος αυτός. Ε, ε, θέλετε να είμαι ειλικρινή ε, μαζί σα, δεν θα μπορέσουμε να τα πράξουμε όλα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα βάλουμε τα δυνατά μα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, λέει ο μιλητή στα αγγλικά, αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μα. Και επομένως, αν θέλουμε τελικά να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου και να έχουμε μία νέα σχέση σε όλες τις διατάσεις, θα πρέπει να λάβουμε περισσότερο χρόνο και να συνεχίσουμε πέρα από τα τέλη του 2020, να εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε με τους Βρετανούς και να διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, θα αναλάβω και μια τελευταία δέσμευση, αν μου επιτρέπει η πρόεδρος Φόντερ Λάιεν και ε, ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια μέθοδο, τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, το διάλογο με το σύνολο των αρμοδίων επιτρόπων και τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Να πω και κάτι τελευταίο στον κύριο Μίκελ Ήβερ, ο οποίος ε, εκφράστηκε πολύ έντονα και μας είπε είμαστε περήφανοι που είμαστε Βρετανοί. Βεβαίως, ε, σεβόμαστε την περηφάνεια αυτή και την κατανοούμε όμως ε, κύριε Βουλευτά. Και εμείς ε, είμαστε εδώ περήφανοι που είμαστε πατριώτες όλοι και δεν θα λάβουμε διδάγματα πατριωτισμού από σας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι για το δικό μας ε, πατριωτισμό, στο δικό μας πατριωτισμό έχουμε και μία πρόσθετη διάσταση. Πιστεύουμε ότι ο πατριωτισμός μας σήμερα και αύριο στον ευριανό κόσμο θα είναι πιο σταθερός, πιο στερεός, γιατί εδώ προσθέτουμε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των Ευρωπαίων και την κοινή δράση των Ευρωπαίων. Ευχαριστούμε κύριε Μπαχνιέ. Και τώρα λοιπόν ε, τελευταίος ε, ομιλητής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Μισελ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώ ε, για τα πολλά και διάφορα μηνύματα που απευθύνατε και εκφράσατε. Πρώτο απ' όλα, το κλίμα ήταν το πρώτο και κύριο διακύβευμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη μερασμένη εβδομάδα. Ε, κατανοώ απολύτω το καθήκον που έχουμε αναλάβει και πρέπει να φέρουμε ει πέρα και την αναγκαιότητα ε, να πετύχουμε του στόχου μα για το 2030, να συμφωνήσουμε για να προετοιμαστούμε και για την επερχόμενη COP25. Να κάνουμε τι απαραίτητε αξιολογήσει για να συνεχίσουμε την πρόοδο σε αυτό το θέμα. Δεύτερο στοιχείο. Πράγματι, πρόκειται για ε, μια πολύ σημαντική απόφαση, απόφαση της περισμένης εβδομάδας που είναι ομόφωνη σε ό,τι αφορά τον στόχο για την κλιματική ουδετερότητα για το 2050 ένα κράτο μέλο, ό,τι αφορά την υλοποίηση και μόνο, θεώρησε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα ακριβώ τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τρίτον, έχετε ανοίξει το θέμα ε, και έχουμε ανοίξει το θέμα ε, του τη οικονομική διάσταση και τη χρηματοδότηση που είναι θεμελιώδε. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια του επόμενου μήνε. Ε, σίγουρα θα έχει να κάνει και με τη συζήτηση για τον επόμενο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Πολλοί το ανέφεραν. Θεωρώ ότι η ισχυρή στάση ε, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για το Green Deal εν ώψη του 2050 είναι μια σαφής εντολή σε διεθνές επίπεδο ε, και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής με την Κίνα την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχή ε, διαξαγωγή αυτής της Συνόδου και προκειμένου από αύριο να, να είμαστε πρωταθλητές ε, σε αυτή τη διαδικασία και προσπάθεια για την ανάπτυξη αλλά και την βιωσιμότητα. Υπάρχει ανυπομονησία και το σέβομαι αλλά δείτε πόσους, πόση διαδρομή και πόσο έδαφο έχουμε καλύψει τους ε, περασμένους μήνες. Μόλις 9 χώρε στι 27 συμμερίζονταν αυτόν τον στόχο της κλιματικής αλλαγή για το 2050 πριν από μερικού μήνες. Πλέον έχουμε ομοφωνία σε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Δεύτερον, το θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Συμμερίζομαι τα όσα ανέφεραν ο κύριος Βέμπερ και άλλοι ευρωβουλευτές. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα Γι' αυτό και πολύ πριν από την ε, Σύνοδο Κορυφή τη περασμένη εβδομάδα, ε, αφιέρωσα πολύ χρόνο για να συναντηθώ με πολλού ε, επικεφαλεί και αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων για να κατανοήσω το διακύβευμα και το πνεύμα συμβασμού. Θεωρώ ότι η πολιτική συνοχή εξαρτάται και από τους πολιτικούς υπευθύνου. γιατί βλέπω εδώ ένα επίπεδο φιλοδοξία, το οποίο είναι ιδιαίτερα νομοποιημένο και δίκαιο έχουμε μαζί μας ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που όλοι έχουν να κάνουν και λογοδοτούν ε, στα εθνικά κοινοβούλια, έχουν να κάνουν με τις ε, πολιτικές πλειοψηφίες που εκπροσωπούν. Επομένω, κατανοώ τη σημασία να υπάρχει μια πολιτική συνοχή και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το μήνυμα που μεταφέρουν οι αρχηγοί. Τέλος, θα ήθελα να σταθώ και στο θέμα της ε, Μάλτας και το κράτος δικαίου. Θέλω να είμαι εξαιρετικά σαφής ε, σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Το κράτο δικαίου είναι, δικαίου είναι μια θεμελιώδης αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δολοφονία μιας δημοσιογράφου σαφώς πρώτα και κύρια είναι ένα δράμα και μια τραγωδία για την οικογένειά τη, ένα, μια ανθρώπινη τραγωδία. Πέραν τούτου όμως είναι και μια βαρύτατη και σοβαρότατη επίθεση στην ελευθερία του τύπου που είναι μια από τι θεμελιώδει ελευθερίε ε, που μα προστατεύουν και μα ενώνουν. Συνεχίζονται οι ε, έρευνες, πρέπει να βασίζονται στο κράτος δικαίου, στην αρχή της, ε, ε, του διαχωρισμού των εξουσιών. Όλοι και ω Ευρωπαίοι ξέρουμε πώς ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Εγώ δεν πρόκειται να υπεκφύγω των δικών μου ευθυνών, κάθε φορά το έχω πει. Είμαι απόλυτα διατεθειμένος να συναντήσω και την οικογένεια της θανού Κάτι τελευταίο για το Brexit. Και θα ήθελα να παραλάβω και εδώ, όπως κάθε φορά, αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με το δημοψήφισμα. Κάθε φορά λοιπόν εκφράζω το σεβασμό μου προ ε, τη θέση και άποψη που πήρε ο Βρετανικό λαό με το δημοψήφισμα. Ε, λυπάμαι για αυτή την απόφαση, αλλά τη σέβομαι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα και όπως είπε και ο κύριος Μπαχνιέ προηγουμένως, με ιδιαίτερη ακρίβεια, ε, ξεκίνησε και πήρε το δρόμο για τα επόμενα βήματα. Ξέρουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε, ξέρουμε που θέλουμε να φτάσουμε και ξέρουμε ότι η διαφάνεια και η ενότητα θα είναι ε, σημεία κλειδί για να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Εμείς θα προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς. Με ηρεμία βέβαια, με ένα πνεύμα αμοψυχίας και ομόνιας, θα ήθελα να πω σε όσους άκουσα προηγουμένως εδώ στην Ολομέλεια, να πω λοιπόν ότι ε, εκείνοι συνεχίζουν να προσβάλλουν ε, παρά να χρησιμοποιούν επιχειρήματα. Ε, να τους πω λοιπόν ότι εμείς δεν πρόκειται να φοβηθούμε εμείς θα ανταπαντήσουμε στι προσβολές με ένα πνεύμα ηρεμία και ομοψυχίας ε, για το κοινό μα μέλλον, για, τις, ε, για τους στενούς δεσμούς που θα μας δένουν με το Μνήμονο Βασίλειο και στο μέλλον. Επαναλαμβάνω την πεποίθηση και τη φιλοδοξία ε, και την εμπιστοσύνη που έχω, την πίστη που έχω σε ό,τι αφορά τις αρχές που θα μας οδηγήσουν στο μέλλον και θα μας επιτρέψουν να φέρουμε εις πέρας και να ελοποιήσουμε το όραμα και τα όνειρα των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Μισελ. Έκλεισε η συζήτηση και θα ακολουθήσει η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Ευχαριστώ.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 Чечне, вообще на Северном Кавказе. Still, there is hope. C'est dramatique.